Ιστάλ που θέλουν να πατάξουν την τρομοκρατία και την ιδεολογικά υποκινούμενη βία να επικρατήσουν. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Επιτροπέ. Έχουμε 7 προτάσεις ψηφίσματος. Θα ψηφίσουμε στις 11.30. Και περάμε στην κατάσταση Καμπότζη. Για ένα λεπτό το λόγο κυρία Γκόμες το πρόβλημα στον αναπτυσσόμενο χώρο με την υφαρπαγή ε, ε, ε, αγροτεμαχίων είναι μεγάλο στην Καμπότζη. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από εθνικές και περιφερειακές αρχές καθώς και επιχειρήσεις. Αυτή η πολιτική που δεν καλύφθηκε από την τελευταία σχετική νομοθεσία παρεμποδίζει την εθνική συμφιλίωση καθώς και τη σταθερότητα στη χώρα, αντίνει ε, ε, τις ανισορροπίες, ε, αυξάνει το εμπόριο όπλων και θέτει την αμφιβόλο την αξιοπιστία της κυβέρνησης. Ασκείται μεγάλη βία κατά των ακτιβιστών και δεν υπάρχει καμία λογοδοσία. Έτσι η κυβέρνηση της Καμπότζης πρέπει να σταματήσει τις εξώσεις από τα αγροτεμάχια και να θεσπίσει ένα νομικό πλαίσιο κατόπιν διαβουλεύσεως με την ε, κοινωνία των πολιτών χορηγώντας αυτούς που έχουν υποστεί έξωση ε, στέγη και γη. Καλούμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παρακολουθήσει εκ του ΣΥΝΕ και στη δραστηριότητα ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην Καμπότζη, διότι ε, δεν πρέπει να μετάσχουν σε αυτές τις καταχρήσεις του νόμου. Ευχαριστούμε, ο κύριος Πρέντα. Για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα να εκφράσω τη λύπη μου για την κατάσταση που παρατηρείται στην Καμπότζη. Ε, οι ακτιβιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ε, έχουν κατηγορηθεί για εγκλήματα. Το 2012, τον Οκτώβρη, στο δικαστήριο της Μνόμ Πένε καταδικάστηκαν και επίσης ένας ραδιοφωνικός σταθμός δέχθη κατηγορίες διότι αναμεταδίδουν επικρίσεις κατά της κυβέρνησης. Αυτό είναι και το μοναδικό τους ατόπιμα. Στην Καμπότζη παρακολουθούνται πολλοί πολίτες από την κυβέρνηση εν ώψη και των κοινοβουλευτικών εκλογών που θα λάβουν χώρα το 2013. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αποστείλει ε, κλιμάκια παρακολούθησης ε, των εκλογών. Η προηγούμενη αποστολή εξέδωσε συστάσεις για την αναβάθμιση του συστήματος. Καλό θα ήταν λοιπόν να εξετάσουμε τα αποτελέσματα και τις συστάσεις και να δούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Ευχαριστούμε κύριο Στάνου και ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Καμπότζη έχει κάνει μεγάλη πρόοδο από τους εκμέρους και την τυραννία. Όμως, με τα έσχατα γεγονότα βλέπουμε ότι ακόμη μένει μακρύς δρόμος. Ε, πολιτικοί κρατούμενοι που ήταν στα χέρια των δυνάμεων ασφαλείας έχουν πεθάνει, έχουν εκτοπιστεί, έχουν χάσει τη γη τους μέσω της νέας νομοθεσίας. Χιλιάδες άνθρωποι δεν υπάρχει διαφάνεια και τρομοκρατούνται οι ακτιβιστές. Οι συντηρητικοί τάζονται υπέρ Τη της Πολιτικής Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Προαγωγή της Δημοκρατίας και των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Καμπότζη πρέπει να μπορούν να διαδηλώνουν χωρίς φόβο, να ψηφίζουν κατά συνείδηση ε, και να μην δέχονται απειλές ε, και ε, το κίνδυνο να χάσουν τα ορθωμάτια τους. Ευχαριστούμε κύριε Τάνο, που ο κύριος Μαστάλκα τώρα παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να υποστηρίξω τις προτάσεις της Ενωμένης Αριστεράς, οι οποίες προτάσεις θεωρούν ότι τα πολιτικά και τα κοινωνικά δικαιώματα είναι άρρηκτα συνεδεμένα μεταξύ τους. Οι τα Ηνωμένα Έθνη ε, δημοσίευσαν στοιχεία ε, οικονομικής φύσεως ε, σύμφωνα με τα οποία η Καμπότζα είναι στην 130 ένατη θέση. Το κατακεφαλή εισόδημα είναι 170 δολάρια μόνο, ενώ στο Βέλγιο είναι πολύ περισσότερα. Στην Καμπότζη το 28% ε, ε, του πληθυσμού ζει με 1,25 δολάρια την ημέρα. Γι' αυτό λοιπόν και εγώ διαρωτώ με τι έκανε άραγε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έτσι ώστε να ε, διατηρούν διατηρηθεί το επίπεδο διαβίωσης των πολιτών. Δεν νομίζω ότι έκανε και πάρα πολλά. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, η πολιτική αναδασμού στην Ευρώπη χαρακτηρίζεται από αυθαιρεσία. 400.000 άνθρωποι έχασαν τη γη στην οποία ζούσαν και εκδιώχθηκαν από αυτή. Ο Πρωθυπουργό Χουνσέν φέτο ανακοίνωσε ότι θα τροποποιηθεί αυτή η άδικη κατανομή γη. Όμως ε, κανείς δεν πιστεύεται την κυβέρνηση. Υπάρχουν ε, ήδη καινούριε ε, περιπτώσεις αδικία και συνεχίζεται η άδικη κατανομή απαλωτριώσεων. Εμεί λοιπόν καλούμε την κυβέρνηση να αλλάξει πορεία και κυρίω να επανεξετάσει το γεγονός ότι έδωσε σε 200 επιχειρήσεις εκτάσει εκτάσεις που θα έπρεπε ίσως να αναθεωρήσει. Όποιος ε, χάνει τη γη στην οποία ζούσε, εκδιώκεται και, ε, και διώκεται. Εμείς υπερασπιζόμαστε όλους τους ακτιβιτές στην Καμπότζη. Υπάρχουν ε, επιχειρήσεις οι οποίες εκμεταλλεύτηκαν αυτή την πολιτική και αυτές οι επιχειρήσεις εξάγουν τα προϊόντα τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν καλείται να καταδικάσει τις ε, παραβιάσεις δικαιωμάτων και αυτό μάλιστα κατά τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο. Sir Watson έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, ο Πρωθυπουργός Χουνσέν έχει την εξουσία 27 χρόνια στην Καμπότζη και η κυβέρνησή του είναι αυταρχική, διεφθαρμένη, ενώ ο κόσμος ζει συνεχώς υπό το φόβο αυθαίρετης κυβερνητικής δράσης. Κάποια η πρόοδος υπήρξε σε μεγάλο βαθμό χάρη και στις προσπάθειες Ευρωπαϊκής Ένωσης η δικαστική εξουσία δεν είναι ανεξάρτητη, οι εκλογές δεν είναι ούτε ελεύθερες ε, ούτε δίκες και μάλιστα την, την προηγούμενη εβδομάδα ο Πρωθυπουργό ε, εξέφερε την ευαρέσκειά του για την πρόθεση των δύο μεγαλύτερων κομμάτων να μποϊκοτάρουν τι εκλογέ. Ενώ η νίκη σε περίπτωση υποκαταρίσματος ε, των εκλογών, η νίκη του θα είναι άνευ αξία και αντικρίσματος, η νίκη του Λουκασέγκο στη Λευκορωσία. Αν δεν έχουμε δίκαιε, ανώθευτε και ελεύθερε εκλογέ, δεν θα πρέπει να, υποστηρι... να υπάρξει διεθνή υποστήριξη για αυτέ. Χαίρομαι για την ανησυχία τη είπα, τη για την κατάσταση στο Μανσανάντο και την Ένωση Δημοκρατών, καθώ και την καταδίκη του περασμένου μήνα κάποιων ακτιβιστών. Ελπίζω να συνεχίσει αμύωτη η πίεση του Συμβουλίου και τη Επιτροπή για την θέση του, του υπεύθυνου της αντιπολίτευσης, του αρχηγού της αντιπολίτευσης Αμνάση, ο κύριος Κέλαμ. Η Καμπότζη έχει σημειώσει κάποια πρόοδο προς τη δημοκρατία, αλλά μας απασχολεί η μοίρα των πολιτών, ιδιαίτερα των ακτιβιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων, γιατί οι ακτιβιστές των δικαιωμάτων ε, αντιμετωπίζονται ως έσχατοι ε, προδότες και μάλιστα πριν από λίγες μέρες καταδικάστηκαν σε φυλάκιση ακτιβιστές ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο δεύτερο ε, λόγο ανησυχία είναι η πολιτική εκχώρηση γεών στην Καμπότζη. Την τελευταία δεκαετία πάνω από μισό εκατομμύρια άνθρωποι εκτοπίστηκαν αναγκαστικά ή έχασαν τη γη τους, τα σπίτια τους με δημεύσεις και παλωτριώσεις. Αυτό οδήγησε και σε συγκρούσεις αλλά και σε όξυση της φτώχειας. Ελπίζω να σταματήσει η παρενόχληση της αντιπολίτευσης και των ακτιβιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Θα θέλαμε να απευθύνουμε έκκληση στην Καμπότζη να τροποποιήσει το εκλογικό σύστημα αναβαθμίζοντα το και φέρνοντα το σε ίσο επίπεδο με τι διεθνεί προδιαγραφέ με βάση τι συστάσει και του ΟΗΕ. Επίση, να σταματήσουν οι αναγκαστικέ εξώσει των ανθρώπων από τα οικόπεδά του και τα γραπτήματά του. Ο κύριο Βάιντερ Χόλτσερ, για ένα λεπτό. Πρόεδρε, το καλοκαίρι που πέρασε εγώ πήγα στην Καμπότζη και έτσι λοιπόν είχα την ευκαιρία με τα ίδια μου τα μάτια να δω ε, και επίσης ε, να διαπιστώσω μόνη μου πως ε, η διαφθορά συμβάλλει στην φτώχεια και πώς ε, όλα αυτά επιβαρύνουν τους ανθρώπους. Η Καμπότζη είναι, αν θέλετε, ο επιμικημένος βραχίωνας ε, της δικής μας της κοινωνίας ε, των πολιτών. Γι' αυτό λοιπόν αξίζει την προσοχή μας. Και μόνο αν επαναφέρουμε τα δημοκρατικά δικαιώματα, μόνο τότε η χώρα θα μπορεί να έχει μέλλον. Με τέτοια μου τα μάτια είδα τις ε, πολιτικές ε, πρωτοβουλίες, ε, πώς αυτές παρεμποδίζονται, πώς δεν υπάρχει ελευθερία και πώς οποιαδήποτε πολιτική δραστηριότητα κινδυνεύει οι επερχόμενες εκλογές που πρέπει να τις παρακολουθήσει εκ του σύνεγγυς η Ευρώπη αυτές μπορούν να αναγνωριστούν ως δημοκρατικές αν ήδη πριν από τις εκλογές υπάρχει η ελευθερία της συγκέντρωσης ε, γιατί μόνο έτσι θα μπορούν να υπάρχουν πραγματικές ελευθερίες. Για τους ε, δημοκράτες ε, και φιλελεύθερους για ένα λεπτό κύριο Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι ένας μακρύτατος ο κατάλογος των ε, εγκλήματων ε, στην Καμπότζη. Διασπάθηση χρήματος, ε, παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά των ακτιβιστών. Έχουμε έναν πανούργο δικτάτορα ο οποίος προσπαθεί να νομιμοποιηθεί. Σήμερα έχουμε και το πρόβλημα των, του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης που έφυγε από την Καμπότζη. Επίσης, ας μην ξεχνάμε ότι δυστυχώς η η κοινωνία των πολιτών, η παγκόσμια κοινωνία ε, φυσικάζει. Είδαμε ότι όταν πήγαμε με τον κύριο Γουτς Βότσον ότι η κατάσταση δεν είναι αρκετά αποτελεσματική, δεν αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά από την ίδια την Επιτροπή. Έτσι λοιπόν εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν γίνει πολλές συζητήσεις για την Καμπότζη και με αρκετό δυναμισμό και θα ήθελα αυτό να επανελειφθεί και σε άλλους θεσμούς. Όσον αφορά τώρα το γκάμα δυνατοτήτων συνεργασίας, νομίζω ότι πρέπει να εξετάσουμε κυρίως στην περίπτωση Σαμ Ράις, ε, ο οποίος πήρε από το ΕΛΚ ένα σημαντικό βραβείο για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ίσως λοιπόν πρέπει να ε, βοηθήσουμε έτσι ώστε να επιστρέψει αυτός και μάλιστα πριν από τις εκλογές. Για τους συντηρητικούς ε, και μεταρρυθμιστές, για ένα λεπτό κυρία Γκέρλινγκ. Ευχαριστώ. Το 2012 η κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Καμπότζη συνεχίζει να επιδεινώνεται. Παραβιάσεις των δικαιωμάτων σε σχέση με τη στέγη και την κατοχή γη συνεχίζονται και επίσης οι ακτιβιστές δέχονται κατηγορίες ε, για παραβιάσεις ανύπαρκτε. Ε, έχουμε πολύ ανησυχητικέ περιπτώσεις σε σχέση με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Ε, στη συνέχεια οι ιδιωτικέ εταιρείε οικειοποιούνται αγροτεμάχια και δεν υπάρχει επαρκής στέγη για τους ανθρώπους. Η αγροβιομηχανία ευθύνεται για πολύ άριθμες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών, υποχρεωτική έξυση, μειωμένη πρόσβαση σε βοσκοτόπια και η φαρπαγή γης από την οποία εξαρτάται και η διαβίωση των ανθρώπων. Το πρόβλημα με τους φυσικούς πόρους της Καμπότζης θα μπορούσε, αν ακολουθούσε μια βιώσιμη ε, και δίκαιη πολιτική, να λύσει τα προβλήματα δικαιώματα των πολιτών τη Καμπότζη, οπότε απευθύνουμε έκκληση προ την κυβέρνηση τη Καμπότζη, να προστατεύσει τα θεμελιώδη δικαιώματα όλων των πολιτών, ούτω ώστε να μπορούν με ειρηνικό τρόπο να εκφράσουν την άποψή του κυρίω σε σχέση με τι επικείμενε εκλογέ. Ευχαριστούμε κυρία Γκέρλινγκ. Ο κύριο Κούκαν, τώρα ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εσχάτως οι ακτιβιστές ε, τρομοκρατήθηκαν από την κυβέρνηση, από τις ε, ιδιωτικές εταιρείες και από την πολιτική ελίτ. Αυτό ε, συνιστά κατάφορη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Ο μόνος Σομάντο και άλλοι ακτιβιστές καταδικάστηκαν σε 20 χρόνια κάθριξη και είναι ξεκάθαρο ότι αυτή η κατεδίκη και οι δίκη καθώς και άλλες πολλές υπακούν σε πολιτική πολιτικές ε, σκοπιμότητες ε, η κατάσταση στην Καμπότζη επιδεινώνεται και θα πρέπει να απελευθερωθούν οι πολιτικοί κρατούμενοι. Αυτό πρέπει να ζητήσουμε. Είμαστε από τους μεγαλύτερους δωρητές ε, ανθρωπιστικής βοήθειας προς την Καμπότζη, οπότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτήν την βοήθεια ως κλίση αφύπνισης για την κατάσταση, κυρίως εν ώψη της επικείμενης συνόδου του Νοεμβρίου σε αυτή τη χώρα. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Κούκαν, ε, σας ευχαριστούμε. Τώρα ένα λεπτό η κυρία Κρέτου, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στο μέτρο που είναι ο βασικός δωρητής ε, προς, της Καμπότζης ε, θα έπρεπε να επικεντρώσει την προσοχή της και την προσπάθεια της ε, στις εκκλήσεις προς την κυβέρνηση για την μεταρρύθμιση του εκλογικού νόμου. Αυτό ζητάει η διεθνή κοινότητα. Ε, η κατάσταση είναι ιδιαίτερα επισφαλής κυρίως ε, με ενόψη των εκλογών που θα διεξαχθούν το 2013. Πρέπει να εξασφαλίσουμε δημοκρατικές εκλογές στην Καμπότζη Καμπότζη ε, και να τηρηθούν και σχετικές συμβάσεις ε, του ΟΗΕ. Έχει ασκηθεί υπέρμετρη βία, μαζικές ε, εξώσεις. Θα πρέπει άμεσα και άνευ όρων να απελευθερωθούν οι πολιτικοί κρατούμενοι, τα μέλη της αντιπολίτευσης, ούτως ώστε να είναι αξιόπιστοι και η αντιπολίτευση. Σας ευχαριστούμε κυρία Κρέτου. Για ένα λεπτό τώρα η κυρία Βίξτρομ παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Επισκέφθηκα τον κύριο Μουσουκού από το Sunrise Party στην Καμπότζη και μου εξήγησαν την κατάσταση για τη γη στην Καμπότζη και ε, δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτές τις εικόνες που είδα. Πάρα πολλές οικογένειες έχασαν και το σπίτι και τη γη τους, ε, το κράτος ε, και οι μεγάλες εταιρείες κατέσχεσαν την, το σπίτι και την γη που δούλευαν αυτοί οι άνθρωποι επί σειρά ετών και δεν έλαβαν καμία καμία αποζημίωση, ε, βρίσκονται χωρίς δικαιώματα, χωρίς καμία ελπίδα. Το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα πάντα εκτός από τα όπλα, ε, επί της αρχής είναι πολύ καλή πρωτοβουλία. Όμως, ε, στην πραγματικότητα είχε ιδιαίτερα ανητικές επιπτώσεις σε σχέση με τη ζάχαρη και άλλα γεωργικά προϊόντα. Αυτές οι γιγάντιες εταιρείες δεσπόζουν στην αγορά και ολόκληρα χωριά, χιλιάδε οικογένειε έχουν μείνει χωρί στέγη για να καλλιεργεί το λένα και περισσότερη ζάχαρη και να εκπληρώνεται η σχετική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε χαίρομαι που μέσα στη συμφωνία συμπεριλαμβάνεται μία έκκληση για να πάψουν αυτέ οι δραστηριότητες ε, και να δώσουμε την ευκαιρία στην αντιπολίτευση, το Sunrise Party, ούτω ώστε να έχει κάποια ελπίδα στι επόμενε εκλογέ. Σα ευχαριστώ. Περνάμε τώρα στο HDI. Για ένα λεπτό, κύριο Σόγκορ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Είναι αλήθεια Πρέπει να γνωρίζουμε ότι τα μέτρα που έλαβαν τα τελευταία χρόνια οι αρχές της Καμπότζης αποτελούν οπισθοδρόμηση. Οι ε, ακτιβιστές φυλακίζονται, η γη κατάσχεται, παράνομα βέβαια, και όλα αυτά καταδεικνύουν πέρα από κάθε αμφιβολία ε, ότι η κυβέρνηση ποδοπατά τα ανθρώπινα δικαιώματα. Γι' αυτό λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει κάτι να κάνει για τη χώρα αυτή. Δεν μπορεί να παραμένει αδρανής ε, και να βλέπει την κατάφορη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η διεθνής κοινότητα οφείλει να μεριμνήσει τον Ιούλιο του 2013 να λάβουν χώρα δημοκρατικές εκλογές στη χώρα. Αλλιώς ε, θα πρέπει να καταγγείλουμε την ε, συμφωνία με την Καμπότζη ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Η κυρία Μακοβέ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Από την Ειρηνευτική Συμφωνία του Παρισίων ε, το 1991 η Καμπότζη προσπάθησε να βελτιώσει την κατάσταση, τη δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δυστυχώς όμως πρόσφατα φαίνεται να έχει παλινδρομήσει στο δρόμο της προς τη δημοκρατία. Γιατί στο ισχύον σύστημα βλέπουμε βία και εκφοβισμό. είμαστε οι περισσότεροι, οι μεγαλύτεροι δωρητές προς την ε, ε, Καμπότζη θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την ε, επιρροή μας και να παροτρύνουμε την Καμπότζη να τροποποιήσει το εκλογικό σύστημα και να δημιουργήσει πρόσφορα περιβάλλον για ελεύθερες και δίκαιες εκλογές. Γιατί μια κυβέρνηση που θα προκύψει από απάτη και τρόμο θα ε, κυβερνήσει με τρόμο και ψέματα. Θα πρέπει επίσης να αποτρέψουμε τη χρήση κατά φίλοι ειρηνικών ακτιβιστών. Θα πρέπει να φροντίσουμε ώστε Καμπότζη να μην εκτραπεί από το δρόμο πρόοδου που έχει ξεκινήσει τα τελευταία χρόνια. Κυρία Γκέριγκερ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Το 1991 η Καμπότζη υπέγραψε τη συνθήκη των Παρισίων αναλαμβάνοντας την ευθύνη να σεβαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μετά από 21 χρόνια ο περιορισμός έκφρασης της ελευθερίας ε, και των ε, μέσων μαζικής ενημέρωσης δυστυχώς αποτελούν καθημερινό πρόβλημα. 13 ε, γυναίκες συνελήθησαν τον περασμένο Μάιο μόνο και μόνο επειδή διαμαρτυρήθηκαν για το νέο οικονομικό σύστημα εκχώρησης των γεών. Πολύ, ένας α, ακτιβιστής και μέλος αντιπολίτευσης καταδικάστηκε σε 20 χρόνια για υποτιθέμενη άσκηση επιρροής και εκφοβισμό προς, μέλη της αντιπολίτευσης. Η κατάσταση των μειονοτήτων επίση είναι ανησυχητική. Θα πρέπει να υπενθυμίσουμε στον κυβέρνηση τη Καμπότζη τι διεθνεί υποσχέσει και δεσμεύσει τη και την εφαρμογή των ψηφισμάτων του ΟΗΕ, εφαρμόζοντα πολιτικέ μεταρρυθμίσει και εξασφάλιση κλίματο για ελεύθερε και δίκαιε εκλογέ, προκειμένου όλοι οι πολίτε να απολαύσουν τα δικαιώματα που απορρέουν από ένα δημοκρατικό καθεστώ. Ευχαριστώ κυρία Όγιουλαντ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε ένας αφιλελεύθερος ε, πολιτικός ε, επισήμανε την κατάσταση στην Καμπότζη και παρόλα αυτά ε, φυλακίστηκε. Είμαι κατά του εκφοβισμού και των συλλήψεων κατά ακτιβιστών ανθρωπίνων δικαιωμάτων μελών αντιπολίτευση αλλά και κατά τη υφαρπαγή γεών στην Καμπότζη. Δεν θα πρέπει η Καμπότζη να υπονομεύσει το δρόμο της προς τη δημοκρατία με τη δίωξη των πολιτικών αντιπάλων. Βέβαια, είναι δύσκολα τα μαθήματα της δημοκρατίας, αλλά αποτελούν αναπόσπαση τμήμα μιας πραγματικά αυθεντικής ε, και δημοκρατικής κοινωνίας. Θα πρέπει ε, επίσης ε, να περάσει τη λιδία λίθο των, τους από τις φόρου τιμή προς τον πρώην βασιλεία. Νομίζω έτσι θα δείξει ότι είναι στο σωστό δρόμο. Κύριος Βλάσεκ, για ένα λεπτό ότι με πρόεδρε, το γεγονός ότι το Κοινοβούλιο επιλαμβάνεται αυτού του θέματος είναι πολύ σημαντικό. Βεβαίως και πρέπει να μιλήσουμε για την πολιτική κατάσταση στην Καμπότζη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας από τους μεγαλύτερους δωρητές και γι' αυτό λοιπόν δεν πρέπει να διασπαθήσουμε αυτήν την οικονομική βοήθεια. Οφείλουμε να αναγκάσουμε την κυβέρνηση στην ε, Καμπότζη να λάβει υπόψη της το ψήφισμα υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Να επιτρέψει στους ανθρώπους να συμμετέχουν ενεργά στην κοινωνία χωρίς αυτό να συνεπάγεται διώξεις. Ευχαριστώ. Η κυρία Κορχόλα για ένα λεπτό. Arvoisa puhemies, kiitos. Kambotsassa valmistaudutaan ensi... Ευχαριστώ, Πρόεδρε στην Καμπότζη προετοιμάζονται για τις εκλογές ε, το 2013 και ως δωρητής η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να υπενθυμίσει την ε, σημασία και το ειδικό βάρος της ελευθερίας έκφρασης. Ε, στις περασμένες εκλογές το κλιμάκιο παρακολούθησης απεφάνθη ότι δεν τηρούνται οι δημοκρατικοί κανόνες κατά τη διεξαγωγή των εκλογών και ζήτησε μεταρρύθμιση της εκλογικής διαδικασίας δημιουργούνται πάρα πολλά προβλήματα διότι με τον περιορισμό της ελευθερίας ε, της έκφρασης η αντιπολίτευση δεν έχει καμία δυνατότητα να κατακρίνει τη διαφθορά Φερρυπίν. Ε, συχνά ε, κρατούνται μυστικά τα στατιστικά στοιχεία. Οι πολίτες ως εκ τούτου δεν μπορούν να μετάσχουν επικοδομητικά στο δημοκρατικό διάλογο. Πρέπει να υπεραμεθεί του κράτους δικαίου η κυβέρνηση της Καμπόντης επιτέλους και να απελευθερώσει τους αντιφρονούντες μετά από την έκθεση σε σχέση με την άσκηση βία και τις αφαίρετες σύλληψη. Ευχαριστούμε. Βερμάγεν, ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Είναι αλήθεια ότι στην Καμπότζα οι δυνάμεις ασφαλείας καταστέλουν βία τα συλλαλητήρια και τις διαδηλώσεις. Πλήττονται κυρίως οι ακτιβιστέ, Έχουμε και ένα κορίτσι 14 ετών το οποίο δολοφονήθηκε από δυνάμεις ασφαλείας και μετά δεν υπήρξε καν έρευνα των συνθήκων δολοφονίας. Ε, άρα δηλαδή είναι αδιαμφισβήτητη η ε, καταστολή των ε, δικαιωμάτων. Οι μικροί γεωργοί χάνουν την γη τους και το αποτέλεσμα είναι ότι γίνονται πολλές εξαγωγές προς την Ευρώπη. Άρα δηλαδή θα πρέπει να πάψει αυτή η εμπορική πολιτική τη στιγμή που η πολιτική που ακολουθείται στη χώρα δεν μας βρίσκει σύμφωνους. Η Επίτροπος έχει το λόγο. Ε, ε, ε, θα ήθελα από πλευρά τη ΕΠΑ τη εκπροσώπου να ευχαριστήσω το Κοινοβούλιο που διοργάνωσε αυτή τη συζήτηση με τι έσχε εξελίξει στην κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Καμπότση τα τελευταία δύο χρόνια. Αυτό κατέστη αναγκαίο. Κατάσταση για του ακτιβιστέ, του δημοσιογράφου και ειρηνικού διαδηλωτέ επιδεινώνεται. Ε, παρακαλώ, ε, ησυχία λέει ο Πρόεδρο. Ε, ε, δεν ετηρούνται βασικά δικαστικά πρότυπα. Το τελευταίο παράδειγμα ήταν ε, η καταδίκη του Μόμ Σενάντο και άλλων ακτιβιστών την 1η Οκτωβρίου σε 20 ετή κάθριξη. Ε, αυτό κατακρίθηκε από την ύπατη εκπρόσωπο, μάλλον την εκπρόσωπό τη και τόνισε ότι δεν υπάρχει ανεξαρτησία στο δικαστικό σύστημα. Η έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Καμπότζη που εξεδόθη τον Ιούλιο 2012 από τον ειδικό εισηγητή, τον καθηγητή Σούριο Σούμπιτη του ΟΗΕ, καθώ και η επιπρόσθετη έκθεση σε σχέση με τι παραχωρήσει Τεμαχίων τη 24 Σεπτεμβρίου επιβεβαίωσαν ε, πόσο σοβαρή είναι η κατάσταση. Ε, μειώνεται το περιθώριο ελιγμών για την κοινωνία των πολιτών ε, ανεξαρτήτως πολιτικού κόμματο για να μπορέσουν να εκφραστούν ελεύθερα και χωρί φόβο. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία διότι επίκυνται τον Ιούλιο του 2013 οι κοινοβουλευτικέ εκλογέ η, η φαρπαγή γεών, αναγκαστικές εξώσεις με έλλειψη σταθερότητας έχουν αναδειχθεί σε μείζον πολιτικό πρόβλημα. Έχουμε καταδείξει ανησυχίε μα σε σχέση με το θέμα των παραχωρήσεων Αιγαίων και σε διάφορα, διάφορες συσκέψεις υψηλού επίπεδου έχουμε θέσει αυτά τα ζητήματα την τελευταία φορά τον Ιούνιο. Τον Απρίλιο ο Επίτροπος Ντεχόχτ επίση συζήτησε αυτό το θέμα επί Μακρόν με τον ομότιμο του τον Πρανσίτ. Ε, ο πρόεδρος Εφανερόμπη από τις 2 μέχρι τις 4 Νοεμβρίου θα μεταβεί στην Καμπότζη και θα έχει την ευκαιρία να συναντήσει τον Πρωθυπουργό Χουν Σενέ, καθώς και τον πρόεδρο της κοινοβουλευτική Συνέλευση. Ο πρόεδρος της Καμπότζη ακόμη, ε, ε, μάλλον συγγνώμη, η Καμπότζη τώρα ε, συνεχίζει τα βήματα προς τον εκδημοκρατισμό και τώρα θεραπεύει τις πληγές του παρελθόντος, όμως υπολείπεται μακρύς δρόμους για να μπορέσει να ανακτήσει το οικονομικό μέρισμα που της αναλογεί. Συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε τις προσπάθειες της Καμπότζης τη δημοκρατική, για τον εκδημοκρατισμό της και 7,5 εκατομμύρια δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως βοήθεια για να ε, υποστηρίξει τη λειτουργία των εκτάκτων δικαστηρίων ε, καθώ ε, και τη Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Από το 2003 και μετά 16 ταμεία έχουν συσταθεί για ένα σύνολο 4,5 εκατομμυρίων βάσει του μέσου για την δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση για να προστατευτούν οι ηθαγενεί, οι πολιτικοί κρατούμενοι και να προαχθούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Επίση, θα αποστείλουμε αποστολή για την παρακολούθηση των κοινοβουλευτικών εκλογών τον Ιούλιο του 2013. Θα συνεχίσουμε συνεχίσουμε να απευθύνουμε εκκλήσει προ την κυβέρνηση, ούτω ώστε να εξασφαλίσει ελεύθερε και δίκαιε εκλογέ, ούτω ώστε και οι υποψήφοι και οι ψηφοφόροι να μπορέσουν να ασκήσουν τα βασικά του δικαιώματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα συνεχίσει να αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συνδέονται με την υφαρπαγή γεών. Σα ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε. Ολοκληρώνεται το σημείο αυτό. Έχω λάβει έξι προτάσεις ψηφίσματος που θα τις ψηφίσουμε εντός ολίγου. Θα κάνουμε τώρα μια πολύ σύντομη διακοπή της Ολομέλειας για να γίνει η ανακοίνωση του βραβευθέντος με το βραβείο Ζαχάροφ και αμέσως μετά θα περάσουμε στις ψηφοφορίες. Ευχαριστώ.